Βίβια, να πιστεύω ότι θα ασχοληθούν επισταμένα με ε, την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο. Έχουμε λοιπόν τρεις ε, προτάσεις ε, ψηφίσματος, καθώς έχει κλείσει η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το πρωί στις 12. Τώρα λοιπόν, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, πάμε στην στα λατωματικά εμφυτεύματα στήθους από σιλικόν της γαλλικής εταιρείας PEP. Ε, Πρόκειται για προφορική ερώτηση ε, προς την Επιτροπή. Και θα ήθελα ευθύς αμέσω να δώσω το λόγο ε, στο συνάδελφο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαστε υποχρεωμένοι να διαπιστώσουμε ότι το θέμα των εφητευμάτων ΠΕΙΠ δεν είναι απλώς ένα θέμα υγειονομικής απάτης σε εθνικό επίπεδο. Βλέπουμε σε ποιο βαθμό δυστυχώς το θέμα αυτό έχει και θα έχει πανευρωπαϊκή και διεθνή ε, διάσταση. Μερικά νούμερα ε, για να καταλάβετε τι λέω. 60, 71 ε, χώρες ε, έχουν αυτά τα εμφυτεύματα να κυκλοφορούν, δηλαδή 400.000 εμφυτεύματα, 40.000 γυναίκες μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, 30.000 στη Γαλλία, 10.000 στην Ισπανία. Η οδηγία για ε, τα ιατρικά βοηθήματα θα αναθεωρηθεί το 2012. Θα πρέπει ε, να λάβουμε τα μέτρα μας, να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας ε, για τα ιατρικά τεχνικά ε, θέματα. Ε, συμφωνώ με τους συναδέλφους Ούλμερ και Φιλίπ Τζουβέ που είναι οι ε, της ερώτησης για το ΕΛΚ που δυστυχώς ε, ζητούν συγγνώμη γιατί απουσιάζουν και θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη τις εξής συστάσεις. Να ενισχύσουμε και να εναρμονίσουμε τις υποχρεώσεις ε, ελέγχου και επιθεωρήσεων. Θα πρέπει η έλεγχη να είναι τακτική απροειδοποιητή αιτήσει σε όλα τα στάδια ε, παραγωγής ενός τέτοιου ιατρικού βοηθήματος. Ε, θα πρέπει επίσης να δούμε πώς εγκρίνονται οι άδειε για τους συγκεκριμένους οργανισμούς ε, και πώς παρακολουθούνται αυτές οι δραστηριότητες στην ευρωπαϊκή αγορά. Επίσης θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στο εξή σημαντικό. Θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των Ευρωπαίων ασθενών και την υποστήριξη στήριξη της καινοτομίας και της έρευνας. Να ε, παντρέψουμε την ασφάλεια με την αποτελεσματικότητα, τη συνέπεια, με την ευελιξία. Ε, δηλαδή, δεν είναι φάρμακα αυτά τα βοηθήματα. Είναι τρεις βασικές διαφορές. Ε, διαφορά από τη φύση τους, διαφορά από τη διάρκεια κυκλοφορία στην αγορά και διαφορά και από τις εγκροές στις αγορές. Το βλέπουμε ότι όταν κυκλοφορούν τέτοια ε, βοηθήματα θα πρέπει να είναι διαφορετική η μεταχείρισή τους από τα φάρμακα. Να μην είναι βαριές οι διαδικασίες αδειοδότης, αλλά να περίπτωση να το ζυγίζουμε και να το σταθμίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, πολύ ωραία. Μακάβεν για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ σχεδόν με όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνει το ψήφισμα που μας έχει κατατεθεί ε, και περιμένω να μας πει ο Επίτροπος κ. Σεντάλη πώς ε, θα γίνει η αναθεώρηση της οδηγίας για τα ιατρικά ε, βοηθήματα. Τι μάθαμε από το σκάνδαλο ΠΥΠ, το οποίο όπως αναφέρθηκε προηγουμένως έπληξε τόσο πολλές γυναίκες στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες. Σήμερα θα σας μιλήσω κάτι, για κάτι ευρύτερο από το ψήφισμα. Πρόκειται για τη δική μου την τροπολογία για τη διαφήμιση. Διότι δεν επιτρέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνεται διαφήμιση για φάρμακα. Όμως επιτρέπουμε ε, κυρίως ε, γυναικεία περιοδικά να ε, δημοσιεύουν τέτοιου είδους εμφυτεύματα και συμβουλεύουν τις γυναίκες πώς μπορούν να βρουν τα καλύτερα. Ε, δύο χώρες, η Γαλλία και το Βέλγιο, δεν το επιτρέπουν. Όμως στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης αυτό είναι φυσιολογικό. Και διερωτώ με κύριε Επίτροπε, μπορούμε να κάνουμε κάτι από αυτού στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί αν δείτε τις ιστοσελίδες αυτών των εταιριών, ε, εκεί ε, προβάλλουν τις ερωτήσεις που τους κάνουν για την εγχείρηση στήθους, τι θα πληρώσει κανείς, πώς θα πάρει δάνειο για να κάνει αυτή την επέμβαση. Πουθενά όμως δεν λέει ότι 30% των γυναικών θα πρέπει να βάλουν νέο εμφύτευμα μέσα σε 10 χρόνια και ότι ε, σχεδόν όλα τα εμφυτεύματα πρέπει να αντικατασταθούν κατά 10 με 15 χρόνια. Δηλαδή στα 32 αν κάνει κανείς κάτι τέτοια επέμβαση σε όλη την υπόλοιπη ζωή του θα πρέπει να βάζει εμφυτεύματα και ξανά εμφυτεύματα. Εγώ λοιπόν είδα τις ιστοσελίδες τριών γνωστών εταιριών και ούτε μία δεν το λέει. Όταν οι άνθρωποι υφίστανται μεγάλες επεμβάσεις, αυτό είναι κίνδυνος για την υγεία τους και αυτό πρέπει να τους το λέμε, να είναι ενημερωμένοι οι ασθενείς. Δεν ξέρω κύριε Επίτροπε τι είδους αρμοδιότητες έχετε. Έχουν με νομοθεσία για τη διαφήμιση των ε, φαρμάκων ε, και πλέον πρέπει να ενημερωθούν οι γυναίκες. Πολλές γυναίκες που ερωτήθηκαν δεν ήξεραν όλα αυτά ότι θα πρέπει να υφίστανται συνεχώς επεμβάσεις κάθε, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ε, ε, Ευχαριστώ η κυρία Λεπάζ για δύο λεπτά. Απουσιάζει. κυρία Όκεν. Øh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πιστεύω ότι για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να ξεκαθαρίσουμε ότι ε, αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ καλύτερες διαδικασίες αδειοδότησης σε σχέση με το παρελθόν. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια και την ε, πρόσβαση σε ανεξάρτητους, απολύτως ανεξάρτητους και αμερόληπτους εμπειρογνώμονες ε, που θα εξετάζουν τα διαθέσιμα δεδομένα με τρόπο ώστε η βιομηχανία να δυνατή να ε, αποκρύψει ε, τα ευρήματα της έρευνας. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θα πρέπει να μπορούν οι άνθρωποι να γνωρίζουν αν υπάρχουν επιβλαβείς συνέπειες, αν έχουν σημειωθεί θετικές αλλαγές ε, σχετικά με οποιοδήποτε ιατροτεχνικό βοήθημα, διότι μην ξεχνούμε ότι υπάρχουν και άλλα βοηθήματα που λειτουργούν αισίως. Ε, Πάντω ε, είναι κέρια σημασίας η διαφάνεια που επιδιώκουμε και ελπιστούμε ότι ο Επίτροπος Νταλή θα ε, λάβει δεόντως υπόψη αυτό το δεδομένο ότι δηλαδή αυτοί που κινδυνεύουν ε, είναι οι πολίτες και όχι η βιομηχανία. Αν λοιπόν υπάρξει παραποίηση, οποιαδήποτε προσπάθεια εξαπάτησης ε, μέσω των δεδομένων, αν υπάρχει έστω και μία υπόνοια για αξιόπινη πράξη, οφείλουμε να προβλέπουμε τις ε, όλοι επιθυμούν ε, την ε, διαφάνεια για τα δεδομένα. Πρέπει να τα επεξεργαζόμαστε, να συνειδητοποιήσουμε πόσο ισχυρό είναι το λόμπινγκ της βιομηχανίας ε, ισχυρίζονται ότι υπονομεύουμε την εμπορική του δράση, τι ε, συνθήκες που θα τους επέτρεπαν να είναι ανταγωνιστικές αυτές οι επιχειρήσεις. Δεχόμαστε δηλαδή μεγάλη πίεση και ελπίζω να αντισταθούμε όλοι σε αυτή την πίεση για να μην ε, υποχωρήσουμε και φτάσουμε στα επίπεδα του ε, Αμερικανικού σχήματος. Ευχαριστώ κυρία Γιανακουδάκη. Δύο λεπτά. Ε, έξι μήνες μετά το σκάνδαλο που βγήκε σε εφημερίδες για τα εμφυτεύματα PIP, ε, αποφάσισε και το Κοινοβούλιο επιτέλους να ασχοληθεί με αυτή την ε, απεχθή περίπτωση ε, κακής ιατρικής πρακτικής. Ο τρίτος μεγαλύτερος προμηθευτής εμφυτευμάτων μπόρεσε για σχεδόν μια δεκαετία να παραβλέψει τον νόμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν από αυτά τα περιστατικά δημόσιας υγείας να καταλάβουμε ότι είναι ζωτική σημασία να εξετάσουμε το σύνολο των δεδομένων προτού καταλήξουμε σε συμπεράσματα αν δηλαδή πρέπει να τροποποιηθεί το σύστημα για την αποφυγή τέτοιων περιστατικών επιπροσθέτω, ε, το σκάνδαλο PIP δεν ε, συνιστά αποτυχία του τωρινού, του ισχύοντο συστήματος συμμόρφωση. Ε, πρόκειται για μια αξιόπινη πράξη όπου τίθεται σε εμπορία ένα προϊόν που δεν πληρεί τα εγκεκριμένα πρότυπα η Επιτροπή ε, θα πρέπει να αναλάβει θετικά μέτρα για να βελτιώσει το νομικό πλαίσιο για τα ιατροτεχνικά βοηθήματα. ζητείτε επίσης ε, πρώτερη αδειοδότηση, δηλαδή πρώτη θέση ε, σε εμπορία. Όμως εδώ ε, υπάρχουν δύο μέτρα και δύο στάθμα σε σχέση με άλλα προϊόντα και άρα δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω. Στην τροπολογία των πρασίνων, παραδείγματο χάρη, ζητούνται ε, ε, αξιολογήσει τη τοξικότητα όλων των βοηθημάτων. Θεωρούμε δηλαδή ότι αν αρχίσουμε να εξετάζουμε ε, του, τις γάζες και τα βήματοδότε, ε, θα βελτιώσουμε ε, την κατάσταση. Παίρνουμε ένα τεράστιο σφυρί δηλαδή για ένα καριδάκι, για να σπάσουμε ένα καριδάκι θα πρέπει να είναι αναλογικά τα μέτρα μα. Το ρυθμιστικό σύστημα ε, για πάνω από 20 χρόνια προστατεύει υπαρκώς τους ασθενείς. Γι' αυτό το λόγο εμείς ε, υποβάλαμε τροπολογίες ε, και αιτήματα για χωριστές και κατατμήματα τμήματα διότι υπάρχουν ανακολουθίες αποφάσεις που παίρνουμε. Σας ευχαριστούμε. Δέχεστε μία μπλε κάρτα, κυρία Γιανακουδάκη. Όχι. Όχι. Catch the Θα τα πείτε στο Catch the Ωραία. Η κυρία Ματίας, ε, τώρα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε αληθεύει ότι πέρασαν έξι μήνες από τότε που συνέβη αυτό το σκάνδαλο ε, ε, των εφητευμάτων PAP. Για πάνω από δέκα χρόνια μια ιδιωτική εταιρεία, όσο απίστευτο και να ακούγεται αυτό, μπόρεσε να διαθέσει στην εμπορία ενθέματα σιλικόνης ε, που θα έπρεπε υποφυσιολογικέ συνθήκε να χρησιμοποιηθούν ω υλικά για τον κατασκευαστικό τομέα και ανταυτού βρίσκονται μέσα στι γυναίκε πολλών δυτικών χωρών. Ε, Εκτιμάται ότι 15.000 γυναίκες επλήττονται από αυτό και ε, πρόκειται μόνο για εκτιμήσεις διότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε αυτή τη διαδικασία. Ξέρουμε ότι αυτό που συνέβη στην ε, περίπτωση αυτή είναι μια απάτη, ένα δίκημα ε, και επιβάλλεται η προσφυγή στη δικαιοσύνη. Τα δικαστήρια θα δώσουν μια λύση για αυτήν την απάτη. Αλλά εμά θα πρέπει να μα ασχολήσει το γενικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο. Δεν καταφέραμε δηλαδή ε, καθ' όλη τη διάρκεια αυτή τη δεκαετία να εντοπίσουμε αυτήν την εγκληματική δράση τη εταιρεία και να την σταματήσουμε. Γι' αυτό σα λέω ότι υπάρχουν ελλείψει. Όλα τα συστήματα που έχουμε για τον εντοπισμό τέτοιων περιστατικών απέτυχαν. Ε, ε, η αρχιοθέτηση των επιστημονικών δεδομένων, το σύστημα εντοπισμού, οι επιθεωρήσει. Πρόκειται για μεγάλη έλλειψη ενημέρωσης και είναι σοβαρό πρόβλημα όχι μόνο σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση αλλά κυρίως διότι πλήττονται χιλιάδες ε, οι γυναίκες ε, κυρίως ε, οι γυναίκες που αναγκάστηκαν να κάνουν και δοκιμές για να συνειδητοποιήσουν τι είδους ένθεμα είχαν μέσα τους είναι πρόβλημα δημόσιας υγείας και δεν μπορούμε να είμαστε τόσο χαλαροί όταν τίθεται τέτοιο ζήτημα δημόσιας υγείας πριν από λίγο καιρό ε, ασχοληθήκαμε με τα ανταλλακτικά των αυτοκινήτων. Λοιπόν, ε, νομίζω ότι αυτό είναι πιο σημαντικό. Το ζήτημα δηλαδή των ιατροτεχνικών ε, βοηθημάτων είναι θετικό που τώρα καταλήξαμε σε αυτό το ψήφισμα, αλλά χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια για να έχουμε και μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλά και κυρώσει, γιατί δυστυχώ αυτό δεν λύνει, οι κυρώσει αυτέ δεν λύνουν το πρόβλημα αυτών των γυναικών που υπέστησαν αυτέ τι επεμβάσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφο Ρώση, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Η συζήτηση για την ψηφοφορία του ψηφίσματο ε, τυχαίνει σε μια πολύ ιδιαίτερη και κατάλληλη στιγμή, γιατί ε, μπορεί πράγματι να γίνει αναθεώρηση των ιατρικών βοηθημάτων. Αυτή η περίπτωση των εμφυτευμάτων δείχνει ότι υπάρχουν πάρα πολλέ λήψει, δεν καλύπτονται οι προδιαγραφέ σε θέματα υγιεινή και ασφάλεια. Εγώ πιστεύω ότι οι προτάσει αναθεώρηση που κατατέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιτροπή από τον κύριο είναι κατάλληλες έτσι ώστε να υπάρχουν μεγαλύτερος έλεγχος των ιατρικών βοηθημάτων και μεγαλύτερη αυστηρότητα από πλευράς αρμόδιων οργανισμών. Συμφωνώ επίσης ότι δεν πρέπει να υπάρχει υπερβολική γραφειοκρατία γιατί για χρόνια ε, παρεμποδίζει την εμφάνιση καινοτόμων προϊόντων. Νομίζω ότι είναι σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρχουν έλεγχοι αποτελεσματικοί και γρήγοροι. Η γυναίκες που ε, βάζουν αυτά τα εμφυτεύματα θα πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους που ενδεχομένω να αντιμετωπίσουν. Να έχουν τη δυνατότητα ε, να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις για να μπορούν να προλάβουν ε, τις διάφορες ε, συνέπειες. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρχει ένα μητρό και να μπορεί να καταφύγει κανείς σε, ε, σε αυτούς που έχουν βάλει αυτά τα εμφυτεύματα έτσι ώστε οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητο να δίδονται πληροφορίες για ελέγχους ή αλλαγές να μπορεί κανείς να το κάνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επίσης είναι απαραίτητο να υπάρχει και μια κάρτα αναγνώρισης των εμφυτευμάτων. Ο χρήστης θα μπορούσε να γνωρίζει όλους τους κινδύνου. Ε, και τους ελέγχους που πρέπει να κάνει μέσα στα χρόνια. Είναι απαραίτητο λοιπόν για να υπάρχει συνεργασία σε κοινωτικό επίπεδο τα κράτη-μέλη να αναλάβουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις για να ελαχιστοποιήσουν την επανάληψη σοβαρών ατυχημάτων όπως έγινε με την περίπτωση των εμφυτευμάτων της εταιρείας PIP. Ο Επίτροπος κύριος Ντάλι έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Τα τελευταία 20 χρόνια το σύστημα ελέγχου των ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων ε, ήταν κάτι που επέτρεψε να κυκλοφορούν αξιόπιστα και ασφαλή βοηθήματα ε, με ε, αξιοπιστία γιατί είναι και σύντομη ζωή αυτών των βοηθημάτων. Το σύστημα είναι αποτελεσματικό, από πλευράς κόστους και φιλικός προς το χρήστη και προς την έρευνα και την καινοτομία. Μήνες πριν την περίπτωση PIP, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεωρούσε την οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα, διότι ε, βρήκαμε ότι ε, χρειαζόταν κάποιες βελτιώσεις. Η περίπτωση PIP είναι πραγματικά ανατριχιαστική. Είναι περίπτωση απάτης δεν ε, ε, αποκαλύφθηκε ε, λόγω της απάτης που έγινε μετά την κυκλοφορία στην αγορά. Το πλαίσιο το κανονιστικό χρειάζεται να προσαρμοστεί για να δώσουμε σύντομη απάντηση στις ανησυχίες των ασθενών και μαζί με το Κοινοβούλιο ταυτοποιήσαμε κάποιες δράσεις που πρέπει να αναλάβουμε σύντομα και μαζί με τα κράτη-μέλη βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Αυτό σημαίνει πιο αυστηρούς ελέγχου της αγοράς για να υπάρχει μεγαλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια και την ιατρική τεχνολογία, ιδιαίτερα βοηθημάτων υψηλού κινδύνου. Γι' αυτό απίθυνα επιστολή στους Υπουργούς Υγείας όλων των κρατών μελών και τους ζητώ την υποστήριξή τους και ε, τα θέτουμε αυτά ε, σε εφαρμογή. Ε, για το πιο μακροπρόθεσμο τώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει μια νομοθεσία ανεξάρτητα από το PIP και θα σημειώσουμε και την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από την υπόθεση αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει μετά τις ενές διακοπές να εγκρίνει πρόσφατα, σύντομα μια νομοθεσία η βελτίωση αυτή θα βοηθήσει να αποτραπούν ε, τέτοιες περιπτώσεις. για αυτήν την παρακολούθηση και ε, τη λειτουργία ε, των οργανισμών και να γίνεται ε, σύμφωνα με τις ε, ίδιες υψηλές προδιαγραφές παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να δοθεί ε, πιο πρωταγωνιστικός ρόλος στις αρμόδιες αρχές ε, και πρώτερη έγκριση αλλά και μετά την έγκριση κυκλοφορία στην αγορά. Για να είναι το σύστημα αποτελεσματικό θα πρέπει να αξιοποιούμε όσο γίνεται καλύτερα τους λίγους εμπειρογνώμονες που υπάρχουν. Γι' αυτό χρειάζεται ένας μηχανισμός ελέγχου πριν την κυκλοφορία στην αγορά για ε, βοηθήματα υψηλού κινδύνου ε, και αναπερίπτωση πολύ σοβαρό έλεγχο. Ο μηχανισμός αυτός θα επιτρέψει σε μια επιτροπή ε, που θα απαρτίζεται από επιρογνώμονες των κρατών μελών να ελέγχει των προτέρων τις αδειοδοτήσεις πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά τα βοηθήματα. Γιατί το κάνουμε αυτό. Θα έχει διπλό όφελος. Πρώτον, θα έχουμε το ίδιο επίπεδο εκτίμησης ειδικά σε σχέση με τα κλινικά στοιχεία και ενιαία αντιμετώπιση. Επιτρέπει στα κράτη-μέλη να ενημερώνονται για προϊόντα που πρόκειται να κυκλοφορήσουν στην αγορά για να κάνουν στοχευμένου ελέγχου. Ο μηχανισμό αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι χρησιμοποιείται πυρογνωμοσύνη και οι πόροι που είναι ε, περιορισμένοι για να έχουμε μεγαλύτερη επαγρύπνηση και παρακολούθηση στην αγορά. Ένα τελευταίο, όχι λιγότερο σημαντικό, θα πρέπει να βελτιωθούν οι απαιτήσει ειχνηλασιμότητα των ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων. Α πούμε, να υπάρχει ενιαία μορφή καταχώρηση και ε, ταυτοποίηση. Μετά την υπόθεση PIP, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ένα έλεγχο, stress test δηλαδή, ε, της νομοθεσίας για να δούμε πώς ε, προσαρμόζεται στη σημερινή πραγματικότητα και πώς θα πρέπει να, ε, να θεωρηθεί όλοι αυτοί οι έλεγχοι έδειξαν ότι ε, θα πρέπει να συμπεριφθούν και νέα μέτρα στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον έλεγχο των εγκεκριμένων ε, οργανισμών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά με την υποχρέωση να γίνονται απροειδοποίητοι έλεγχοι στους παρασκευαστές ε, και να αλλάζουν οι ελεγκτές, να μην είναι οι ίδιοι οι ε, εθνικέ αρχές θα ενημερώνονται για τα αρνητικά αποτελέσματα τέτοιων ελέγχων. Επίσης θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να ενισχυθεί η αναφορά επεισοδίων ε, και προβλημάτων από το υγειονομικό προσωπικό και από τους ασθενείς. Θα πρέπει για παράδειγμα ε, να υπάρχει και μία κάρτα εμφυτεύματος που να ενημερώνει σωστά την κάθε και να γνωρίζει τι γίνεται και έτσι η διαφάνεια της αγοράς θα μπορέσει να ενισχυθεί, ε, να έχουν το δικαίωμα για σε σωστή πληροφόρηση όλοι οι ενεχόμενοι. Όχι μόνο για το κόστος όπως είπε η κυρία Μακάβεν και το όφελος, αλλά τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Ε, πόσο διαρκεί το εμφύτευμα και ποιες είναι οι συνέπειες μιας τέτοιας επέμβασης ή οποιοδήποτε άλλο βοηθήματος. Δεν μιλώ μόνο για τα εμφυτεύματα θέματα. Υπάρχουν και άλλα πολύ σημαντικά βοηθήματα ε, που χρησιμοποιούνται. Και θα πρέπει να γνωρίζει ο καθένας ε, τις συνέπειες ε, των πράξεών του και των χρήσεων τέτοιων βοηθημάτων. Επίσης, επειδή ορισμένοι πιστεύουν ότι όταν κάνουν μια επέμβαση είναι άπαξ και τελείωσε και είναι εντάξει για όλη τους τη ζωή. Δεν συμβαίνει αυτό σε πολλές περιπτώσεις και ε, αυτό θα πρέπει ε, να προβάλλεται διαρκώς και να το γνωρίζουν οι ασθενείς και οι ε, καταναλωτές. Ότι αυτό που προτείνουμε, αυτή η κάρτα λοιπόν εμφυτεύματος θα πρέπει να δίδεται σε κάθε ασθενή για οποιαδήποτε διαδικασία που αφορά τέτοια βοηθήματα και τέτοια εμφυτεύματα. Έτσι θα έχουν γνώση και επίγνωση οι ε, ασθενείς. Ε, αγαπητοί ευρωβουλευτές, Πιστεύω ότι τα μέτρα που ήδη προβλέπονται σε συνδυασμό με τα πρόσθετα μέτρα που θεωρήθηκαν απαραίτητα μετά το αποτέλεσμα των ελέγχων ε, κοπόσεως θα βελτιώσουν το σύστημα, θα ευνοήσουν την καινοτομία και θα εξασφαλίσουν ότι θα κυκλοφορούν στην αγορά της Ευρώπης μόνο ασφαλή ε, βοηθήματα προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Σημείωσα αυτό που ανέφερε η κυρία Οκονή και θα συμπεριλάβουμε όλες τις ανησυχίες και όσα μας επισημάνατε. Σας ευχαριστώ. Eh, Εκ μέρους ε, του ΕΛΚ, ο κύριος Γκαρντίνη για 1,5 λεπτό. Κυρία, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Επίτροπο γιατί είπε πραγματικά πολύ σημαντικά θέματα με τα οποία συμφωνώ και εγώ και όπως είπε και, ο, και εκείνος ε, θεωρώ πραγματικά ε, αποτρόπαιο το γεγονός ότι σε ένα από τα κράτη-μέλη μας βιώσαμε αυτό που ανέφερε προηγουμένως η συνάδελφος. Είναι όμως σαφές ότι το σκάνδαλο αυτό κατέδειξε την αναγκαιότητα να προσαρμοστεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όσον αφορά τα ιατροτεχνικά βοηθήματα. Ε, η ε, απάτη αυτή κατέδειξε τα κενά τα οποία έχουμε εντοπίσει μέχρι τώρα, τα έχουμε επισημάνει στην Ολομέλεια, τα είπε και ο Επίτροπος και γι' αυτό δεν θέλω στο σύντομο διάστημα που έχω στη διάθεσή μου να αναφερθώ σε όλα αυτά. Είναι σωστό να γίνουν τα απαραίτητα έτσι ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατόν στους ε, πολίτες μας. Εγώ όμως ε, πιστεύω ότι το σκάνδαλο αυτό που μας δίδαξε πάρα πολλά, το σκάνδαλο αυτό θα μπορούσε επίσης να αποτελεί ρίσμα για να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός. Προηγουμένως ο συνάδελφος είπε ότι η ενημέρωση που γίνεται προς τους ασθενείς είναι ελιπέστατη. Ε, αναφέρονται μόνο τα θετικά. Τους λένε ότι υπάρχει ένα είδος μόνιμης αιωνιότητας και ομορφιάς, δεν υπάρχουν εμφυτεύματα ε, τα οποία να μην έχουν κανένα απολύτως κίνδυνο και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν οι ασθενείς. Όταν μιλάμε για αισθητικές παρεμβάσεις θα πρέπει να ενημερώνονται οι κοπέλες γιατί συνήθως είναι πολύ νέες κοπέλες αυτές οι οποίες ε, κάνουν αυτές τις επεμβάσεις να ενημερώνονται για τους κινδύνους. Εγώ λοιπόν ε, θεωρώ, είμαι πεπισμένη για όλα αυτά και θα έλεγα να συνεργαστούμε γιατί δεν έχουμε ε, πολύ χρόνο. Θα έπρεπε να έχουμε αποφασίσει ήδη εχθές. λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, είχαμε άλλα σκάνδαλα, τώρα έχουμε το σκάνδαλα των εμφυτευμάτων η δυσλειτουργία αυτό δείχνει τη δυσλειτουργία της ε, προστασίας ε, των ασθενών. Έχουμε ένα σκάνδαλο που διέρχεσε πολλά χρόνια και δεν τιμωρήθηκε κανείς. 500.000 εμφυτεύματα έχουν τοποθετηθεί στον κόσμο. Χρειάστηκε να αφαιρεθούν πάρα πολλά. Είχαμε πολλές περιπτώσεις διαπιστωμένου καρκίνου και ατελείωτες μηνύσεις που υποβλήθηκαν. Όλα αυτά μας σοκάρουν. Παρόλες τις ε, του MDA και των πολλών παραπώνων και καταγγελιών για τα εμφυτεύματα αυτά που κατατέθηκαν στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία. Πόσοι αρμόδιες υπηρεσίες παράβλεψαν αυτή την τεράστια πάτη. Αυτό μας κάνει να σκεφτούμε μια βελτίωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου των Εμφυτευμάτων όπως μόλις το εξηγήσατε και εσείς. Κύριε Επίτροπε, σήμερα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο σύστημα που θα μας επιτρέψει να αποφύγουμε τα σκάνδαλα. Πρέπει να χτίσουμε ένα νέο σύστημα. Προβλέπετε αυτή η νέα νομοθεσία για το φθινόπωρο και ως ε, συνσυντάκτης αυτής της πρότασης είμαι ικανοποιημένος. Αλλά κύριε Επίτροπε, φαίνεται ότι θέλετε να λάβετε υπόψη πάρα πολλές από τις ανησυχία μας, έτσι όπως περιέχονται στο σχετικό ψήφισμα. Γιατί λοιπόν να προβλέψετε μια εξαίρεση απαράδεκτη για πάρα πολλούς βουλευτές που είναι παρόντες σήμερα εδώ. Γιατί να μην θελήσετε τη δημιουργία μιας ειδική άδεια κυκλοφορία στην αγορά για τα αμφιτέματα της κατηγορίας 3 που είναι και τα πιο επικίνδυνα. Μπορείτε να μου εξηγήσετε ποια είναι η θέση σας κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ. Τους φιλελεύθερους η κυρία Μπιλμπάου. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τι προβλέπετε μέσα στα πλαίσια των εμφυτευμάτων ώστε να μην είναι επικίνδυνα. Πολλά μάθαμε από τη μεγάλη κρίση των εμφυτευμάτων ΠΕΙΠΕ. Μας ενδιαφέρει ανταλλαγή στοιχείων και συστήματα προειδοποίησης για να βελτιωθούν και οι δοκιμές σε σχέση με τα εμφυτεύματα αυτά χρειάζεται ένα σύστημα κυρώσεων έτσι ώστε οι προμηθευτές επικίνδυνων ουσιών να μην ε, την χάνουν πάρα πολύ ε, στεναρή, στεναρού ελέγχου. Όλα θα πρέπει να ελεγχθούν με δυνατή φωνή και επειδή προσπαθούμε να, να λύσουμε και να βοηθήσουμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, θα πρέπει να το βοηθήσουμε σε όλους τους τομείς. Τα προϊόντα ΠΕΙΠΕ δεν έτυχαν αυστηρού ελεγχού και κυκλοφόρησαν ε, τα εμφυτεύματα ΠΕΙΠΕ παρόλα αυτά στην αγορά παρά τον ασθενή έλεγχο. Είμαι σίγουρη ότι με τον έλεγχο αυτό που θα γίνει δεν θα ξανασυμβεί μια τέτοια ιστορία, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου και εποπτείας για να μπορέσουμε, να μπορέσουμε ώστε να τηρηθεί αυτό το, το ψήφισμα, αυτή η αρχή με βάση αυτό το ψήφισμα. Η αρχή δηλαδή του στενού ελέγχου. Κάτσε αι τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση. Μιλάμε για, όταν μιλάμε για αυτό το συγκεκριμένο σκάνδαλο πρέπει να παραδεχθούμε ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία βοήθησε πάρα πολύ τους ασθενείς μου αρέσει λοιπόν η ισορροπημένη προσέγγιση του, του Επιτρόπου σχετικά με τη βελτίωση της κατάστασης και για την παράχραβο 7 θέλω να, ε, δεν θέλω, πρέπει να εμποδίσουμε την καινοτομία σε επίπεδο βιομηχανίας. Πρέπει να βρούμε μια σωστή ισορροπία ανάμεσα τι είναι καλό για τους ασθενείς και πώς θα βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής εκείνων που χρειάζονται ιατροτεχνικά βοηθήματα και ε, σε μιλώντας για κάτι διαφορετικό μετά από αυτά μας είπε η κυρία Μακαβάν είχαμε μια συζήτηση για την, ε, τον ακροατηριασμό των γεννητικών οργάνων των ε, γυναικών τώρα μιλάμε για προσθετικά και αμφιτε... προσθετικές παρεμβάσεις και εμφυτεύματα. Παρόλο που δεν συνδέονται τα δύο, οι δύο συζητήσεις, είναι ενδιαφέρον ότι έλαβαν χώρα και οι δύο απόψε. Και αυτό που θέλουν να παρατηρήσουν και άνθρωποι που έχουν εμφυτεύματα ε, στο ισχύο ή στο στήθος, για να, για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους πρέπει αυτό να το επιτρέψουμε χωρίς να πνίγουμε την καινοτομία. Το θέμα των, ε, ε, των εμφυτευμάτων στήθους είναι επίσης ένα θέμα σοβαρό και το, το οποίο θα χρειαστεί να συζητηθεί με κάποια άλλη ευκαιρία. Ο κύριος Ρέγνερ. Κυρία Ρέγνερ, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, θέλω να αναφερθώ σε έναν κανονισμό που ολοκληρώνεται ο κανονισμός πρέπει να τύχει περαιτέρω επεξεργασίας. Μιλάω για το Βρυξέλλες 1, για την δικαστική δικαιοδοσία και την εκτέλεση ε, αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις. Στην Αυστρία υπάρχουν 60 θύματα ε, από τα ελαττωματικά εμφυτεύματα που δεν ενημερώθηκαν. Οι οργανώσεις καταναλωτών τους είπαν να υποβάλουν μήνυση και δεν μπόρεσαν γιατί υπήρχε κενό στην νομοθεσία. Ε, μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση των θυμάτων αν δώσουμε ε, δυνατότητα στις οργανώσεις καταναλωτών να ε, αξιοποιούν τη βελτιωμένη νομοθεσία. Η αποκλειστική δικαιοδοσία ε, πρέπει να τύχει περαιτέρω επεξεργασία στον κανονισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Επίτροπε, μιλάμε για ένα μεγάλο σκάνδαλο ως προς τη χρήση των ΠΙΠ που ήταν εμφυτεύματα στήθους από σιλικόνη βιομηχανικής χρήσης γιατί οι γυναίκες δεν μπορούν να ξέρουν ποια, πώς έχουν αυτά τα εμφυτεύματα και τι είδος σιλικόνη χρησιμοποιείται. Υπάρχουν πολλά νομικά κενά και θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος και ένα σύστημα προειδοποίησης γιατί τα εμφυτεύματα αυτά αφορούν 30.000 γυναίκες Ευρωπαίες και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτά τα προϊόντα ε, είναι ασύμβατα με την υγεία. Θα πρέπει λοιπόν οι γυναίκες να είναι καλά πληροφορημένες και παράλληλα να μην διατρέχουν κανένα κίνδυνο. Διότι οι γυναίκες που βάζουν αυτά τα εμφυτεύματα θα ήθελαν να μην διατρέχουν κινδύνους ως προς την υγεία τους. Ταραμπέλα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπο, μπορεί να σκεφτούμε γιατί υπήρξε διαφορία από πλευράς δημοσίων αρχών. Θέλουν τα θύματα να τους προταθούν συγκεκριμένες λύσεις. Δεν, οπωσδήποτε αυτά που έγιναν δεν είναι τέλεια. Οι επεμβάσεις που έγιναν από τους χειρουργούς για να αφαιρέσουν τα ε, ε, εμφυτεύματα, τα εμφυτεύματα, τα ελαττωματικά, δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και μετά από την ερώτηση που σας επέβαλε στις 13 Ιανουαρίου μου είπατε η, συμπερίληψη ιατρο, ε, ορισμένων ιατροτεχνικών επεμβάσεων για αισθητικούς λόγους είναι αποδεκτή σε αυτό το πλαίσιο Κύριε Επίτροπε, τι θα γίνει σχετικά με τα ιατροτεχνικά βοηθήματα και ποια θα είναι το πεδίο εφαρμογής αυτής της νομοθεσίας στα καλοπιστικά ε, βοηθήματα. Και θα ήθελα να ξέρω πότε ακριβώς θα συμβεί αυτό. Κυρία Κάντεμπαχ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Σήμερα μιλάμε για ιατροτεχνολογικά βοηθήματα και χρειάζονται αυστηρές διαδικασίες εγκρισής, ελέγχου και ενημέρωσης. Τα εμφυτεύματα είναι ένα μεγάλο κομμάτι ε, της αισθητική χειρουργικής πέρα από τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα. Μιλάμε για ένα, μια αγορά 7 εκατομμυρίων. Ε, θα ήθελα να συμφωνήσω με τον κύριο Μακάβερν και να πω ότι θα πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι στον τομέα της υγείας. Πολλές Ευρωπαίες, γιατί γυναίκες είναι κυρίως, ε, έχουν μια διαστρεβλωμένη εικόνα για τον εαυτό τους και νομίζουν ότι με αυτά τα εμφυτεύματα θα γίνουν πιο γυναίκες. Και το 22% των νέων πρωτίστως των γυναικών στην Ευρώπη ε, έχουν ε, τέτοια προβλήματα με την ταυτότητά τους τα οποία βεβαίως δημιουργούνται και από τις εικόνες των ΜΜΕ. Ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων αυτών πιστεύουν ότι με χειρουργικές επεμβάσεις θα αποκτήσουν πάλι αυτοεκτίμηση. Νομίζω λοιπόν ότι για λόγους πρόληψης ε, της υγείας ε, θα πρέπει να ε, δράσουμε και όχι να... Σινκλέρ. Η κυρία Σανκλέρ. Όλα αυτά προέκυψαν για την έλλειψη ρύθμισης από πλευράς γαλλικών αρχών για ορισμένους τομείς. Το Ιούνιο του 2000 οι ρυθμιστές για τα ιατρικά θέματα δημοσίευσαν στο διαδίκτυο τα προβλήματα που υπάρχουν στη Γαλλία για τα αμφιτεύματα. Οι γαλλικές αρχές δεν έδωσαν ιδιαίτερη σημασία το θέμα. Χρειάζονται λοιπόν βασικές αλλαγές σε ό,τι αφορά τη χρήση ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων. Η Γαλλία πρέπει να προβεί σε ελέγχους, διότι πάρα πολλές γυναίκες εξακολουθούν να υποφέρουν για την εμέλεια των γαλλικών αρχών Χρειάζεται μεγαλύτερη επικοινωνία με τους χειρουργούς και τους ασθενείς. Οι εταιρείε πρέπει να ελέγχονται και να τους επιβάλλονται κυρώσεις όταν δεν συμμορφώνονται. Ε, Ευχαριστούμε. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος ε, Νταλή, ο Επίτροπος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τα σχόλιά σας επί αυτού του πολύ σημαντικού ε, ζητήματος. Όλοι συμφωνούμε ότι η υγεία του ασθενούς είναι το πρώτο στο μέλημά μας. Και αυτό ακριβώς κάνουμε όταν λέμε ότι πρέπει να έχουμε ένα ευέλικτο σύστημα έτσι ώστε να προβάλλουμε την καινοτομία το ταχύτερο δυνατό στους ε, ασθενείς διότι έχει μεγάλη σημασία για την υγεία τους. Θα πρέπει να μπορούμε να χρησιμοποιούμε καινοτόμα προϊόντα εν ευθέτω χρόνο και την καινοτομία την προωθούμε στην Ευρώπη τρία χρόνια πριν από τους ομολόγους Αμερικανούς. Αυτό είναι ένα ευεργέτημα προς τους ασθενείς που δεν μπορούμε να αμελήσουμε. Γι' αυτό όταν με ρώτησε ο κύριος Παρνιό γιατί δεν προωθώ την αδειοδότηση ελεύθερης εμπορίας του απαντώ ότι δεν το κάνω διότι θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα προέγκρισης εμείς. Ε, Προσπαθούμε ώστε το σύστημα να λειτουργεί ακόμα καλύτερα έτσι ώστε να είναι αρμόδια όλα τα σώματα στη διαδικασία διοδότησης. Και αυτό είναι το πακέτο το οποίο θα υποβάλουμε στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Μετά από το καλοκαίρι. Και κύριε Ταραμπέλα, αυτή θα είναι η έκβαση του θέματος. Είχαμε προωθήσει διαβουλεύσεις και δοκιμές και θα υποβάλουμε μία επίσημη πρόταση γύρω στο Σεπτέμβριο. Όταν λοιπόν μιλάμε για διαδικασία αδειοδότησης, λέμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε με την ευελιξία που έχουμε στην Ευρώπη, να ενισχύσουμε τη διαδικασία μέσω αρμοδιοτήτων και τα κράτη-μέλη και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή τη διαδικασία και ας έχουμε μία Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ε, Ευρωπαϊκής Εμβέλειας, έτσι ώστε να είμαστε συνεκτικοί και συνεπείς, γιατί η υπόθεση των εμφυτευμάτων ΠΙΠ δεν έχει σχέση με αδειοδοτήσεις. Πρόκειται για ε, μία απάτη η οποία θα μπορούσε να αφορά μία ε, οποιαδήποτε κατάσταση σε μία εύρωστη οικονομία δεν έχει σχέση με την νομοθεσία, αλλά με τον τρόπο που εφαρμόστηκε. Διότι σημασία έχουν οι έλεγχοι στις αγορές μετά από τις αδειοδοτήσεις. Όπως είπαν μερικοί από εσά, οι αρμόδιες αρχές, τα κράτη-μέλη, δεν προέβησαν σε ελέγχους, σταμάτησαν τους ελέγχους ως προς τα εμφυτεύματα αυτά στις χώρες και αυτό εδώ είναι το λάθος. Όλοι οι έλεγχοι που διενεργήθησαν από τις αρχές ειδοποίησης είχαν μία περίοδο δύο μηνών για τη διαδικασία έγκαιρης προειδοποίησης. και θεώρησαν ότι αυτό ισχύει στο νομικό μας σύστημα, κάτι το οποίο δεν ισχύει και αυτό είπα και στους υπουργούς. Θεωρούμε ότι αυτοί οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται εκ των προτέρων. Controls today. We Να μην είναι δηλαδή προγραμματισμένοι οι έλεγχοι, αλλά να γίνονται ευνηδιαστικά και δειγματοληπτικά, χωρίς προειδοποίηση. Θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια, όχι μόνο στις πληροφορίες που δίνονται, αλλά να υπάρχει διαφάνεια ως προς την επαγρύπνηση, δηλαδή όλα τα συμβάντα μέσα στα πλαίσια του ιατρικού κλάδου εμφυτευμάτων, θα πρέπει να επανορθωθεί και να υπάρχει μια τράπεζα δεδομένων που να διαθέτει όλα αυτά τα στοιχεία έτσι ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε τις κατάλληλες δραστηριότητες όπως ως προς την ίχνη λασιμότητα που προτείναμε και που θα προτείνουμε και σήμερα. Αυτή είναι μια επίσης πολύ βασική πτυχή, η ίχνη λασιμότητα όλων αυτών των ε, ιατρικών μέσων, ιδιαίτερα των πλέον επικινδύνων. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε και τον Σεπτέμβριο θα προβάλλουμε μία εύρωστη πρόταση έτσι ώστε να προωθήσουμε την ασφάλεια, θέματα ασφάλειας χωρίς να αντιδράσουμε υπερβολικά ως προς ένα συμβάν. Χωρίς να κάνουμε κάτι εκεί που δεν υπάρχει λόγος να γίνει. Το θέμα της απάτης των εμφυτευμάτων PIP δεν αφορούσε την αδειοδότηση αλλά τους ελέγχους της αγοράς. Και εδώ θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να γίνονται ε, συγκεκριμένοι και δραστήριοι έλεγχοι της αγοράς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο. Ανακοινώνω ότι λάβαμε μία πρόταση ψηφίσματος. Η συζήτηση έκλεισε και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12 το μεσημέρι. Η επόμενη συνεδρίαση προβλέπεται αύριο 14